να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για το θέμα. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αρμόδια για το θέμα, ενημέρωσε τον Πρόεδρο ότι μετά την απόφαση του εφετείου του Βουκουρεστίου να αποσύρει μια ε, προσφυγή που έγινε για πλήρη ακύρωση της απόφασης από το Δικαστήριο του Βουκαστηρίου στη διαδικασία μιας αστικής υπόθεσης υπέρ του κυρίου Βίκτορ Μποστινό